για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώ και του καθεστώτο που εφαρμόζεται στο ελληνικό προσωπικό των κοινοτήτων αυτών. Επίση, έχουμε τι εκθέσει Γουαλτιέρη και Σουριάν σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού για το τμήμα υπαριθμών 2, το τμήμα 3 και το τμήμα 10. Το τελευταίο αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπατε εκπρόσωπε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε και κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, οι οποίοι βρίσκονται καθοδόν, έχουν μείνει μάλλον στην κυκλοφοριακή κίνηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνουμε το τελικό βήμα μιας συναρπαστικής νομοθετικής και διοργανικής περιπέτειας τετραμερούς διαλόγου, δηλαδή την θέσπιση μιας αποτελεσματικής, φιλόδοξης και στραμμένης προς το μέλλον Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης το κείμενο που έχουμε με τροποποίηση του κανονισμού προσωπικού, του νοσονομικού κανονισμού και τον διορθωτικό προπολογισμό που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο, αποτελούν την ε, έκβαση, επιτυχή έκβαση μηνών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Όλων ενωμένων σε ένα κοινό στόχο, το πώς δηλαδή θα οργανωθεί ο τρόπος με τον οποίο ακούγεται η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα εισακούεται αυτή η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Εμείς από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύνε μας στην περιπέτεια αυτή, στη διαπραγμάτευση αυτή με κύριο γνώμονα την, στη δράση αυτής της υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως την επικράτηση του κοινοτικού συμφέροντος, του κοινού συμφέροντος. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν θα διεξαχθεί σήμερα η συζήτηση και έτσι περαιτέρω με αυτό το πνεύμα προσμένουμε με δημονία την, θέση σε, την επίσημη θέση σε λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως το Δεκέμβριο του 2010, μόλις ένα χρόνο μετά τη θέση εφαρμογή της συνθήκης, θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Ξεκινάμε ακούγοντα πρώτα του συζητητέ μα. Η κυρία Γκρέσλιν, είναι η πρώτη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Σεύσκοφης, κύριε Επίτροπε Λεβαντόφσκη, κυρία Αντιπρόεδρε, ε, αν είπατε εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσει την ανάληψη δράσεως αυτή η υπηρεσία, η ΕΕΔ, μέχρι